και είναι προς το συμφέρον όλων μας να έχουμε έναν πιο αξιόπιστο τρόπο ε, υλοποίησης του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ώρα αυτή των ερωτήσεων. Θα ε, συναντηθούμε και πάλι τον επόμενο μήνα την ώρα των ερωτήσεων και στις συζητήσεις αύριο. Ευχαριστώ πολύ που απαντήσατε. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφοι για τις ερωτήσεις που θέσατε. Ε, Το επόμενο θέμα είναι προφορικές ερωτήσεις. Οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Ε, ε, Καταρχήν ο κύριος Νικόλαος Κούντης. Και πού μας πήγε λοιπόν αυτές που μας υποβάθμισε, junk, junk. Τέσσερις, κατηγορίες κάτω μας πήγανε. Δηλαδή πήγαμε στο κάτω γκρουπ. Β, β. Β κάτι ήμασταν, τρία. Λοιπόν, δεν τίποτα αυτό. Ε, τι λένε αυτοί πια, δεν αλλάζει τίποτα, έχουμε Λοιπόν, σα χαιρετώ. Γεια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE <laughs> Έλα μωρέ, γιατί ήρθες. Μας δύο. μας λίγο με την Κατέρινη. αξιολόγηση Moody's προσπάθησε να δημιουργήσει ξανά αρνητικό κλίμα για την ελληνική οικονομία και το ευρώ με μια ομή κερδοσκοπική παρέμβαση υποβαθμίζοντας χωρίς ουσιαστική αιτιολόγηση την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας κατά τέσσερις βαθμίδες. η moody's είναι μία από τις τρεις αμερικάνικες ιδιωτικές εταιρείες που επίσημα αναγνωρίζει η ευρωπαϊκή ένωση ω του αξιολογητές των οικονομιών των κρατών μελών. παρά το γεγονό ότι καταγγέλλεται από όλου οικονομικού, πολιτικού και θεσμικού παράγοντε σε ευρώπη και αμερική για τι τεράστιε ευθύνε που έχει για την πρόσφατη κρίση. πιο συγκεκριμένα είναι αυτή η εταιρεία που καταγγέλθηκε από πρώην αναλυτέ τη στο αμερικάνικο κογκρέσο ότι εξαναγκάστηκαν από του προϊσταμένου του να κάνουν θετικέ εκτιμήσει για τοξικά χρεόγραφα. είναι αυτή η εταιρεία που καταγγέλλεται από δεκάδε επιχειρήσει ότι εκβίαζε μέσω των αξιολογήσεων με σκοπό την καταβολή αμοιβών. είναι αυτή η εταιρεία που δέχτηκε μαζί με την υπόλοιπη αγία τριάδα των οίκων αξιολόγησης S&P και Fitch δεκάδες μηνύσεις από δήμους περιφέρειες και πολιτείες των ηνωμένων πολιτειών που παραπλανήθηκαν και υποχρεώθηκαν να επενδύσουν και να χάσουν εκατομμύρια δολάρια. είναι αυτή η εταιρεία που καταγγέλλεται από πολλά ασφαλιστικά ταμεία ότι έχασαν τις επενδύσεις λόγω εσφαλμένων αξιολογήσεων μόνο στην περίπτωση του ασφαλιστικού ταμείου της πολιτείας του οχάιο χάθηκαν 450 εκατομμύρια δολάρια. επειδή όλα τα παραπάνω είναι γνωστά κύριε πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι επειδή δεν είναι δυνατόν να αξιολογούν τις ευρωπαϊκές οικονομίες αμερικάνικες ιδιωτικές και ιδιωτελείς εταιρείες θα έπρεπε αυτό το έργο να το έχει αναλάβει ένας δημόσιος δημοκρατικά ελεγχόμενος φορέας ο οποίος να μην έχει καμία σύνδεση με ιδιωτικά συμφέροντα. αντί όμως για αυτά κύριε, ε, ακόμα και σήμερα είμαστε στο σημείο να ακούμε από την κομισιόν να κολυσιεργεί με συνέπεια η μαφία των κερδοσκόπων να συνεχίζει και να εκβιάζει και να κατευθύνει την οικονομική πολιτική σε βάρος των εργαζομένων και των πολιτών των χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης. κύριοι συνάδελφοι κύριε πρόεδρε νομίζω ότι το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο επιτέλους πρέπει να αναλάβει τις δικές του ευθύνες να παρέμβει να απαιτήσει από την ευρωπαϊκή επιτροπή και το συμβούλιο αφού λάβουν υπόψη το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο να νομοθετήσουν άμεσα ώστε να θέσουν τέρμα σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Thank you. Thank you very much. Ο κύριος Πιτέλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι. Με αυτή την προφορική ερώτηση η ομάδα των Σοσιαλιστών και των Δημοκρατών θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή όλων στα θέματα των οργανισμών rating ε, για να μας πει η Κομισιόν ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις λαμβάνοντας υπόψη ε, το, την επιθυμία μας να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή, ένα ευρωπαϊκό οργανισμό rating ε, σημείο το οποίο θεωρώ ότι αποκτά μεγαλύτερη σημασία λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις του Προέδρου κ. Μπαρόζο οι εταιρείε αυτές κατάφεραν αυτό το οποίο θα θεωρούσαμε mission impossible. Δηλαδή, ήδη από το 2008, όταν ξεκίνησε η οικονομική κρίση, όταν χρεοκόπησαν, χρεοκόπησαν οι Lehman Brothers, ε, και μετά συνεχίσαμε και με τις ε, και μετά συνεχίσαμε και με, την, με τα προβλήματα στην Ελλάδα λοιπόν εκεί ε, θεώρησαν ότι θα έπρεπε να ε, επικυρώσουν τα ταξικά προϊόντα και τότε και τώρα θεωρούν ότι υποστηρίζουν ε, την, ε, την έξοδο από την κρίση ε, δημιουργώντας ε, περισσότερα προβλήματα και υποβαθμίζοντας ε, την, την, την οικονομία της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Ιταλίας. Λοιπόν, δεν θεωρώ ότι όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο οφείλονται σε αυτές τις, αυτές τις εταιρείες που, που κάνουν το rating, αλλά παρόλα αυτά οτιδήποτε οτιδήποτε, όποια πέστρα και αν σηκώσει και όποιο πρόβλημα παρουσιάζεται στην, στην οικονομία, στην παγκόσμια οικονομία, αυτοί οι οργανισμοί αξιολόγηση τη πιστοληπτική ικανότητα είναι από κάτω. Επομένω, ε, και το συζητήσαμε και με τον, το ασχοληθήκαμε με τον συνάδελφο Κοζέσο όταν εξετάζαμε τον κανονισμό που αφορούσε του οργανισμού αξιολόγηση, ε, Λοιπόν, τώρα θα πρέπει να ρίξουμε ένα φως σε αυτή την σκανδαλώδη ε, κατάσταση των, ε, της δημιουργίας του, του ολιγοπολίου στην κατάσταση αυτή, στην τομέα αυτό. Θα πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Πριν επιδεινωθεί η κατάσταση, θα πρέπει από τα λόγια να περάσουμε στις πράξεις. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε έναν Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αξιολόγησης και θα πρέπει να σκεφτούμε τον ρόλο που θα μπορούσαν να παίξουν τα ανεξάρτητα ελεκτικά συνέδρια όταν αξιολογούν αξιολογούν ε, τα κρατικά ομόλογα και τα, αυτοί θα πρέπει να αξιολογούν ε, τα κρατικά ομόλογα και όχι οι ιδιωτικοί οργανισμοί ο Σαρκοζή και η Μέρκελ ζητήσαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσουν ε, περισσότερα μέτρα έτσι ώστε να οργανωθεί καλύτερα η, αγορά που, όπου λειτουργούν οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ε, ικανότητας. Και τελικά, παρά την θέληση, των, ε, ε, την θέληση του Σαρκοζή και της Μέρκελ, τελικά είναι οι ίδιες οι κυβερνήσεις που καθυστερούν τη δημιουργία αυτού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού. Επομένως, την την επιστολή κύριε Σα Νικολά και κύριε Άγγελα δεν θα πρέπει να στείλετε στον Αμπαρόζο αλλά στον, στους εαυτούς σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πιτέλα. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Μπαγνιέ που ήρθε και είναι μαζί μας σήμερα. Ε, σας καλωσορίζω με μία μικρή καθυστέρηση, αλλά τέλος πάντων παρόλα αυτά ε, χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Ο κύριος Γκοζές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπη, αγαπητές συνάδελφοι. Ε, το θέμα του Οργανισμού Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας ε, υιοθέτησε και το Κοινοβούλιο μας και στο τέλος της προηγούμενης θητείας ε, και θα ήθελα να υπενθυμίσω την, τα, την θέληση και της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου με την υιοθέτηση του προηγούμενου κανονισμού. Σήμερα θέτουμε ξανά το ερώτημα ε, για να δούμε ποιο ρόλο έπαιξαν οι οργανισμοί αυτοί στην ε, διάρκεια της κρίσης. Ε, μπορούμε να τους κατηγορήσουμε ότι δεν είδαν την κρίση να έρχεται. Μπορούμε να τους κατηγορήσουμε ότι γιατί οι βαθμολογίες αυτές, οι αξιολογήσεις αυτές ήταν κάπως κειμενόμενες. Το γεγονός ότι δεν, δεν αξιολόγησαν σωστά τα, το, τα Όμω, Όμως οι επενδυτέ οι οποίοι επενδύουν και οι οποίοι φέρουν χρήματα θα πρέπει να γνωρίζουν του κινδύνους ή τι δυσκολίε που μπορεί να προκύψουν. Όπω επίση θα πρέπει να ξέρουν του καλου βαθμού. Εκεί που η κατάσταση είναι κάπω πιο διφορούμενη είναι όταν οι βαθμοί αυτοί αν θέλετε ε, χρησιμεύουν ε, στι τράπεζε έτσι ώστε να καθορίσουμε ε, την, τους ίδιου πόρους που πρέπει να έχουν οι τράπεζε σαν αντιστάθμισμα των επενδύσεων θέσεών τους και ε, η κατάσταση το 2009 δεν μας ε, βοηθάει να δημιουργήσουμε μια σαφή εικόνα όσον αφορά την επίβλεψη και τη λειτουργία των οργανισμών αξιολόγησης. Το πρόβλημα είναι, είναι ε, σωστά να, κάνει, να υπάρχει βαθμολογία, αλλά είναι νόμιμο να διαδίδεται και να, η αξιολόγηση αυτή με τον τρόπο που την διαδίδουν οι οργανισμοί αξιολόγησης. Υπάρχει ένα κείμενο, Πρόεδρε, για την εφαρμογή της, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού μηχανισμού αξιολόγησης μέσα στα πλαίσια του νέου δημοσιονομικού κανονισμού και εκεί θα πρέπει να δοθούν ε, απαντήσεις ε, καταρχάς όσον αφορά τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους διάφορους οργανισμούς ε, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι το να πούμε ότι θα δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός οργανισμός έστω και αν είναι δημόσιος θα μας λύσει τα προβλήματα έστω και αν ένας οργανισμός αξιολόγηση ευρωπαϊκός βαθμολογεί πιο ευγενικά από ότι οι ιδιωτικοί οργανισμοί. Το πρόβλημα είναι πώ κυκλοφορούν αυτές, αυτοί αυτέ οι βαθμολογίε, αν θέλετε. Υπάρχουν βαθμολογίες για τις ιδιωτικέ επιχειρήσεις και βαθμολογίες που αφορούν τα κρατικά ομόλογα. Τι γίνεται με τα κρατικά ομόλογα. Η αρχή η οποία θα πρέπει να αναλάβει και το θέλει σε αυτό το κοινοβούλιο να επιβλέψει τους οργανισμούς που θα παρεμβαίνουν στην Ευρώπη είναι η ΕΣΜΑ που είναι η νέα υπηρεσία που δημιουργείται και πιστεύω ότι στις αρμοδιότητες που θα αναλάβει αυτή η νέα υπηρεσία θα πρέπει να μην είναι μόνο η επίβλεψη των οργανισμών αλλά όσον αφορά τα κρατικά ομόλογα να προβλέπει και ε, μία διαδικασία που θα επιτρέπει ε, τον μηχανισμό χωρίς να εφαρμόζει κυρώσεις αλλά να ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί αξιολόγησης ε, κυκλοφορούν τις βαθμούς που αφορούν τα κρατικά ομόλογα. Δεν μπορούμε να δούμε να, να επαναλαμβάνεται 15 λεπτά πληκρίσουν οι αγορέ να υποβαθμίζει ένα τέτοιο οργανισμό σε μια χώρα που δεν μπορεί πλέον να κάνει τίποτα. Επομένω, θα πρέπει να δημιουργήσουμε έναν προληπτικό μηχανισμό ο οποίο θα αναγκάσει του οργανισμού αξιολόγηση σε σύντομο χρονικό διάστημα, ε, λίγο πολύ βέβαια, ε, να ε, ενημερώνει για τη βαθμολογία που πρόκειται να βάλει, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι οι κανονικές διαδικασίες έχουν γίνει σεβαστές, αλλά και να είμαστε σίγουροι ότι οι συνθήκες διάδοσης των πληροφοριών αυτών να μην επηρεάζει την μοίρα των κρατικών ομολόγων. Διότι δεν μπορούμε τα κράτη να αντιμετωπίζουμε με, την, με τον ίδιο τρόπο όπως και με κάποια ιδιωτική επιχείρηση. Βέβαια, υπάρχουν χώρες που έχουν ανεξάρτητα ελεκτικά συνέδρια και άλλες ε, όχι. Τέλος πάντων, Πρόεδρε, ε, θα πρέπει να δούμε πώς θα πρέπει να ε, βελτιώσουμε την λειτουργία αυτών των οργανισμών, τον τρόπο διάδοση των αποφάσεών τους και την, τον ανταγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γκουλά, την επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. έρχεστε από μια χώρα όπου όταν υπάρχει αξιολόγηση σκεφτόμαστε αμέσως τον οδηγό για τα εστιατόρια, τον οδηγό Μισλά. Η αλήθεια είναι ότι συμφωνώ απολύτως με τον Σοπολ σε αυτά που είπε για την αξιολόγηση και τους οργανισμούς αξιολόγησης. Δεν είναι αυτή υπεύθυνη για όλα τα κακά. Πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο και με ποιες προϋποθέσεις εργάζονται και αξιολογούν. Πρόκειται για οργανισμούς που έχουν σημαντική ε, δύναμη και αρμοδιότητες και ο Ζων Πολ είπε κάτι το οποίο συμφωνώ ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της αξιολόγησης ενός ιδιωτικού ε, οργανισμού είτε ε, ενός δημόσιου χρέους. Πώς, παραδείγματος χάρη, ένα κράτος διαχειρίζεται τα ελλείμματά του, αν υπάρχει διαφάνεια και εάν υπάρχει σχέση συνεργασίας ή εμπιστοσύνη μεταξύ αυτού ο οποίος αξιολογεί και του αξιολογούμενου. Το Κοινοβούλιο είχε κάνει κάποιες προτάσεις στην τελευταία θητεία του βάσει της έκθεσης του Ζων Και θα πρέπει να ξαναδούμε αυτές τις προτάσεις καθότι ήδη έχουμε υιοθετήσει κάποιες πολύ σωστές θέσεις. Και εγώ θεωρώ ότι δεν είναι προτεραιότητα να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός οργανισμός αξιολόγησης. Και πρέπει καταρχήν να διαπιστώσουμε, και αυτό είναι πολύ πιο επίγον, το κατά πόσο οι έλεγχοι που γίνονται είναι αξιόπιστοι. Είμαι εισηγήτρια όσον αφορά το πακέτο για την επιτήρηση των χρηματαγορών. Και θα ήθελα εδώ να κάνω μια έκκληση προς τα κράτη-μέλη. Ξέρω ότι η Προεδρία δεν είναι αυτή τη στιγμή παρούσα, αλλά ξέρω κύριε Επίτροπε ότι κάνετε σοβαρές προσπάθειες για να προχωρήσει το θέμα αυτό. Δεν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κατακρίνοντας τους οργανισμούς αξιολόγησης και την ίδια ώρα να μην αφήνουμε την ανεξάρτητη αρχή που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εδώ στην Ευρώπη να την παρεμποδίζουν και να μην θέλουν να προχωρήσει. Θεωρώ ότι ο έλεγχος των οργανισμών αξιολόγησης είναι πολύ σημαντικός. Η επιτήρηση από μια ευρωπαϊκή αρχή των ε, χρηματαγορών, και όλων των οργανισμών που λειτουργούν με αδιάφανο τρόπο στις ε, χρηματαχωρές της Ευρώπης και τις παγκόσμιες χρηματαχωρές. Θεωρούμε ότι ο τρόπος που αξιολογούνται κάποιες υπηρεσίες θα πρέπει να υπακούν σε κανόνες διαφάνειας και τήρησης κάποιων αρχών. Καλούμε λοιπόν όλα τα κράτη-μέλη να μην εμποδίσουν την ε, δημιουργία αυτής της ανεξάρτητης αρχής να μην εμποδίσουν την προώθηση αυτού του πακέτου μέτρων για την επιτήρηση των χρηματαγορών, γιατί όλοι πιστεύω επιθυμούμε αυστηρότερο έλεγχο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κυρία Γκουλάρ και θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο, στον κύριο Μπαρνιέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα ειλικρινά καταρχήν να ευχαριστήσω τις πολιτικές ομάδες που πήραν την ε, πρωτοβουλία να υποβάλουν ε, αυτή την ομάδα των ερωτημάτων. Τους ε, κύριους Χουντή, Γκουλάρ και λοιπά, και τον κύριο Γκοζές. Και ε, θα ήθελα να σας πω και εγώ την γνώμη μου. Θα δείτε πόσο αποφασιστικός είμαι για ένα τέτοιο θέμα το οποίο άπτεται και της κρίσης της διαφάνειας διαφάνεια την οποία αξίζουν και οι πολίτες μας και οι επιχειρήσεις μας. Στις 20 Απριλίου ε, συζήτησα και ε, σχολίασα και πάλι το θέμα των εικόνων που ε, είναι σημαντική για τη λειτουργία της αγοράς γενικότερα και των χρηματοπιστωτικών αγορών ειδικότερα. Για να αξιολογήσει κανείς την ποιότητα ενός προϊόντος, μιας επιχείρησης ή και ενός ε, κράτους, ε, ε, ε, πώς το κάνει. Σίγουρα δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον πυρετό σπάζοντας το θερμόμετρο. Θα πρέπει να δούμε αν το θερμόμετρο λειτουργεί σωστά. Για την ακρίβεια θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε πολλά διαφορετικά θερμόμετρα για να επιβεβαιώνει το ένα το άλλο. Και η άποψή μου είναι ότι έχουμε πολλά να πούμε για τη λειτουργία του θερμομέτρου. οι οίκοι αξιολόγηση παίζουν ένα ρόλο για την αξιολόγηση των, των κρατών και των επιχειρήσεων. Και όπως είπε και ο Χουντής, η λειτουργία των οίκων αξιολόγηση δεν ήταν πάντοτε επιθυμητή, πολλές φορές μάλιστα ήταν και πολύ κακή. Γι' αυτό και το G20, η ομάδα G20 πήρε την απόφαση να αρχίσει να εποπτεύει τους οίκους αξιολόγησης και να ακολουθήσει μια πολιτική καλύτερης διακυβέρνησης. Η Κομισιόν ανέλαβε αμέσως τις ευθύνες της και έθεσε ως προτεραιότητα τη ρύθμιση της λειτουργίας των οίκων αξιολόγησης τα τελευταία αυτά δύο χρόνια. Από το 2009 ξεκινήσαμε, υιοθετήσαμε τον, τον κανονισμό για τους οίκους αξιολόγησης αμέσως μετά την πτώχευση του Lehman Brothers ε, και με αυτόν τον τρόπο προσπαθήσαμε να ε, λύσουμε τα προβλήματα των οίκων αξιολόγηση σε, κάποιο βαθμό. Ε, απαιτήσαμε την εγγραφή του σε Μητρό και επιβάλλουμε συγκεκριμένους κανόνες στη λειτουργία τους προκειμένου να αποφύγουμε συγκρούσεις συμφερόντων, να βελτιώσουμε τη μεθοδολογία της βαθμολόγησης και να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί οι οίκοι δρούν με πιο διαφανή τρόπο. Είμαι σίγουρος ότι αυτοί οι καινούργιοι κανόνες θα βελτιώσουν ε, την ανεξαρτησία των οίκων, ε, την ακαιρεότητα της δράσης τους, την διαφάνεια και την ποιότητα της βαθμολόγησης, της αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης και της βαθμολόγησης των, του δημοσίου χρέους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν από δύο εβδομάδες και αυτή την δεύτερη φάση, στις 2 Ιουνίου, η Κομισιόν μετά από πρότασή μου υιοθέτησε μια πρόταση τροποποίησης του κανονισμού ε, έτσι ώστε ε, να ανατεθεί στην μελλοντική Ευρωπαϊκή Αρχή ε, Αγορών, Χρηματοπιστωτικών Αγορών, τους ελέγχους. Αυτή είναι η ΕΣΜΑ. Η ΕΣΜΑ, και συμφωνώ με την κυρία Γκουλάρ, θα πρέπει να αναλάβει. Και θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα αξιόπιστο συμβιβασμό ανάμεσα στο σύμβολο και το Κοινοβούλιο επί του, των συμπερασμάτων της έκθεσης της ομάδας Λαροζιέρ. Από την, ε, θα πρέπει μέχρι τέλος του χρόνου να τα έχουμε καταφέρει και κάνουμε μια έκκληση και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο να κάνουν προσπάθειες συμβασμού. Εμείς από πλευρά της Κομισιόν θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενθαρρύνουμε αυτό το συμβασμό. Να είναι μεριά, για να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τη διαφάνεια και να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των οίκων αξιολόγηση, εισάγαμε μία ε, διάταξη για την πρόσβαση σε διαρθρωμένες πληροφορίες για όλους τους οίκους αξιολόγησης. Δηλαδή, α, ε, όταν μία, ένας οίκος αξιολόγησης λαμβάνει κάποιες πληροφορίες για την αξιολόγηση κάποιου συγκεκριμένου προϊόντος κλπ. Ε, και οι άλλοι οίκοι αξιολόγηση θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες. Αυτό όμως δεν αρκεί. Ε, είναι αναγνωρίζεται πλέον και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο ότι οι αδυναμίες, οι σημερινές αδυναμίες της διαδικασίας αξιολόγησης δεν έχουν ακόμα ε, ε, ε, διορθωθεί. Και συμφωνώ με τον κύριο Χουντή στην ανάλυση του. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο. Θα ξεκινήσουμε ένα προβληματισμό για την συνολική αρχιτεκτονική και το ρόλο των εικοναξιολόγηση. Γι' αυτό, ε, κύριε Πιτέλα, του επόμενου ε, μήνε θα γίνει η αντικειμενική ανάλυση, πολύ λεπτομερή αντικειμενική ανάλυση τη λειτουργία αυτών των εικοναξιολόγηση. εν ώψη υπό το φως μάλλον της καινούργιας νομοθεσίας, παρόλο ότι θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το Δεκέμβρη για να δούμε τα πλήρη αποτελέσματα αυτής της καινούργιας νομοθεσίας. Ε, αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη αγορά είναι ε, σε πολύ λίγα χέρια δεν υπάρχει υπαρκή ανταγωνισμό μεταξύ οίκων αξιολόγηση ε, και αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Υπάρχει συγκέντρωση. Η Κομισιόν σκέφτεται μέχρι και διαρθρωτικά μέτρα, για παράδειγμα τη δημιουργία ενό ευρωπαϊκού ανεξάρτητου οίκου αξιολόγηση πιστοληπτική ικανότητα. Ε, ιδιαίτερα Κατά την άποψή μου θα είναι χρήσιμη αυτή η υπηρεσία, αυτός ο οίκος θα είναι χρήσιμος για την αξιολόγηση του δημοσίου χρέους, δηλαδή της πιστοληπτικής ικανότητας κρατών. Επίσης σκεφτόμαστε την πρόσθετη συμμετοχή ε, κρατικών αρχών στην ε, ε, αξιολόγηση. Τώρα, για το δημόσιο χρέος μια και μιλάμε για την ε, Ελλάδα. Ε, τα κράτη πρέπει να υπόκειται σε ιδιαίτερου κανόνε, η αξιολόγηση των θα πρέπει να υπόκειται σε ιδιαίτερου κανόνε για να είμαστε σίγουροι ότι γίνεται σωστά. Ε, δεν υπάρχουν εναλλακτικά κριτήρια για την αξιοπιστία επίσης, για την φερεγγιότητα μιας επένδυσης. Χρειάζεται και εκεί να παρέμβουμε. Όλα αυτά είναι τα αντικείμενα πάνω στα οποία θα εργαστούμε στο μέλλον. Δεν αποφεύγουμε κανένα δύσκολο θέμα. Το Σεπτέμβριο θα είμαστε έτοιμοι να εκδώσουμε τις πρώτες κατευθύνσεις ραμές ενώ παράλληλα θα εξετάζουμε και το θέμα του ελέγχου και της διαφάνειας ε, για, για τα παράγωγα προϊόντα και τις ε, ακάλυπτες πωλήσει. Ε, οπότε ε, θα έχουμε ολοκληρώσει αυτή μας τη δουλειά, ελπίζουμε, μέχρι τις αρχές του 2011 και θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε διότι όλα αυτά δεν είναι αρκετά, θα πρέπει να πάμε ακόμη πιο μακριά για να εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια και την, ε, να καταπολύσουμε τις συγκρούσεις συμφερόντων. Θέλουμε οι οίκοι να είναι πιο πολυάριθμοι, να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα και να τους κάνουμε πιο αξιόπιστους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων, ο κύριος Σάντσες προσθέτει για τρία λεπτά. Οι οίκοι αξιολόγηση δεν κατάφεραν να προβλέψουν ε, τις, ε, την κρίση ε, των στεγαστικών δανείων ούτε την κατάρρευση της Lehman Brothers. Ο κανονισμός που εθετήθηκε τον Απρίλιο του 2009 προβλέπει διαφάνεια, επιβάλλει ευρωπαϊκή εποπτεία στους οίκους αξιολόγησης και προσπαθεί να βελτιώσει την αξιοπιστία τους προσπαθώντας ταυτόχρονα να αποφύγει και τις, τις συγκρούσεις συμφερόντων. Και η καινούργια ίδια Κομισιόν συνεχίζει προ την ίδια κατεύθυνση. Νομίζω ότι εμεί εδώ από το Κοινοβούλιο θα συνεισφέρουμε έτσι ώστε ο 1η Ιανουαρίου 2011 να ξεκινήσει η εποπτεία και μάλιστα θα συνεργαστούμε με την Κομισιόν προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα πιο αυστηρό νομοθετικό ε, ρυθμιστικό πλαίσιο. Ε, η οίκη ε, ε, έχουν αυτή τη στιγμή ε, ε, μεθόδους ε, και κανόνες ε, που χρειάζονται ρύθμιση. Πολλές φορές ιδρούν σαν πυρομανείς που αυξάνουν τα προβλήματα αντί να τα μειώσουν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αποφασίσει να πάψει να χρησιμοποιεί ε, τις, ε, τα πορίσματά τους σε σχέση με την αξιολόγηση του δημοσίου χρέους. Ε, αυτό κάτι δείχνει. Το ερώτημα είναι αν αυτή τη στιγμή και οι αξιολόγηση μπορούν να είναι αντικειμενικοί, ιδιαίτερα στην αξιολόγηση του δημοσίου χρέου. Και οι ερωτήσει που τίθενται ε, έχουν ένα διαρθρωτικό, δομικό χαρακτήρα. Δεν ξέρουμε αν αυτή η οίκη αξιολόγηση συμβαδίζουν με το δημοκρατικό χαρακτήρα του πολιτευματό μα. Διότι πολλέ ε, φορέ. Ε, ε, έρχονται σε αντίθεση, η λειτουργία τους έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα των εργαζομένων, των ταξιούχων κλπ. Ε, είναι συμβατό μια ιδιωτική εταιρεία να αξιολογεί κράτη. Είναι δυνατόν αυτή η αξιολόγηση να γίνεται με βάση ε, χρηματοδότηση που προέρχεται από τους αξιολογούμενους. Το Γερουσία των ΗΠΑ εξετάζει ήδη αυτά τα ερωτήματα και πρέπει και εμείς να τα εξετάσουμε είναι θέματα που έχουν σχέση με την βιωσιμότητα και την ευθύνη. Ε, είναι δυνατόν να παραμείνουμε αδιάφοροι ε, στις δεσμεύσεις των κρατών και των διεθνών οργανισμών. Μπορούμε να αγνοήσουμε τις ε, οδυνηρές συνέπειες που προκαλεί η λειτουργία τους διεθνείς αγορές. Μπορούμε να αγνοήσουμε ε, τις, ε, την ανάγκη ρύθμισης ε, του πλαισίου λειτουργίας τους. Μπορούν αυτές, αυτοί οι αξιολόγηση με ελάχιστο έλεγχο να διατηρήσουν την εξουσία που έχουν στις οικονομίες μας. Είναι δυνατόν να υπόκεινται μόνο σε εσωτερικούς ελέγχους. Δεν θα έπρεπε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα αξιολόγησης. Δεν θα έπρεπε να έχουμε να επιφυλάξουμε καινούριο ρόλο στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες ή ενδεχομένως να ε, δημιουργήσουμε και ένα παγκόσμιο οίκο αξιολόγησης. Ευχαριστώ. Η επόμενη, ομιλή... η επομενη ομιλητρια ομιλήτρια κυρία Μπούλς, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Επίτροπε, πριν από λίγο καιρό Ακούστηκαν φωνές ε, για το ότι οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας δεν θα έπρεπε να υποβαθμίσουν ε, τα κρατικά ομόλογα της Ελλάδας. Δείτε τι κάνουν στο ευρώ. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να πούμε για να δείξουμε την σύγκρουση συμφερόντων που θα, θα δημιουργούνταν εάν οι ίδιες οι χώρες έπρεπε να αξιολογήσουν την πιστοληπτική τους ικανότητα ε, Ακούσαμε ότι η υποβάθμιση από, το Moody's, από την Moody's ε, δεν, ήταν σε καλή, δεν ήρθε σε καλή χρονική συγκυρία. Καταλαβαίνω τα προβλήματα, αλλά το πρόβλημα μου είναι τι θέλετε. Θέλετε ε, αξιολογήσει, οι οποίε να, να βολεύουν, τι, πού να βιολεύουν, να βολεύουν τις ιδιωτικές τράπεζες, να βολεύουν τις ε, δημόσιες τράπεζες. Οι αξιολογήσεις είναι ε, καλές φαίνεται και βολεύουν αυτούς που, να βιολευουν να βολευουν τις ιδιωτικε τραπεζες να βολευουν τις δημοσιες τραπεζες οι αξιολογησεις ειναι καλες φαινεται και βολευουν αυτους που την, που παίρνουν κάποιες αποφασει βιαστικε θα τις χαρακτήριζα. Το πρόβλημα είναι πώς θα, βρούμε κάποιες εγγυήσεις, πώς θα έχουμε ε, συγκεκριμένες προφυλάξεις αν θέλετε. Έχουμε κάποιο δρόμο ακόμα να διανύσουμε όσον αφορά την ακαιρεότητα και την ε, ασφάλεια. Το ένα όμως ε, είναι ότι οι αρχές ε, συνετής διακυβέρνησης ε, θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλους τους οργανισμούς. Είτε πρόκειται για ιδιωτικούς οργανισμούς, είτε πρόκειται για την ΕΣΜΑ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριος Γκίγκολτ για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μπανιέ, σας ευχαριστώ πολύ και για τη χρήση της γερμανικής γλώσσας. Η κρίση μέσα στην οποία βρισκόμαστε δείχνει ότι υπάρχει πληθώρα προβλημάτων. Και μάλιστα θα ήθελα να πω ότι ιδιαίτερα κάποιες πτυχές επηρεάζουν σήμερα πολύ την κατάσταση. Οι οργανισμοί αξιολόγησης λειτουργούν σήμερα με έναν τρόπο θα έλεγα μονοπωλιακό, σαν να είναι οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να αξιολογήσουν τους κινδύνους. Υπάρχουν ε, την ίδια ώρα και κάποιοι άλλοι που αξιολογούν και ίσως με διαφορετικό τρόπο και με διαφορετική οπτική γωνιά. Γι' αυτό ακριβώς και θα ήταν κατά την άποψή μου πιο λογικό να διευρύνουμε το φάσμα αυτών που αξιολογούν και να υπάρχουν ίσως και περισσότεροι και πιο πολυάριθμοι αξιολογητές. Ποια είναι τα κίνητρα τελικά. Και νομίζω ότι αυτό μέχρι τώρα δεν συζητήθηκε. Αυτοί οι οργανισμοί αξιολόγησης ουσιαστικά λειτουργούν με έναν τρόπο που θυμίζει κατά κάποιο τρόπο τους ε, καθηγητές που αξιολογούν τον μαθητή ή τον φοιτητή και κατόπιν υπάρχει και ένα, αν θέλετε, χρηματικό αντάλλαγμα το οποίο πολλές φορές ξεχνάμε στην περίπτωση των οργανισμών αξιολόγησης είναι σαν ο καθηγητής να αξιολογεί, να βαθμολογεί τους μαθητές του και να περιμένει κατόπιν και ένα χρηματικό αντάλλαγμα από αυτόν ο οποίος ζήτησε τη βαθμολόγηση. Καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχει κάποιο πρόβλημα και πολλές φορές όταν πρόκειται για δημόσια ελλείμματα και για δανεισμό κρατών βλέπουμε ότι αυτοί που ζητούν την αξιολόγηση είναι ιδιωτικοί οργανισμοί, ιδιωτικοί φορείς. Εδώ λοιπόν πολλές φορές υπάρχει ένα δεύτερο πρόβλημα. Μία δημόσια αρχή, ένας δημόσιος οργανισμός θα μπορούσε ενδεχομένως εδώ να παίξει έναν λίγο διαφορετικό τρόπο, να αντικατασταθεί το ολιγοπόλιο των οργανισμών αξιολόγησης των σημερινών με μια δημόσια επιχείρηση, ένα δημόσιο οργανισμό. Αυτό προτείνουν οι αριστεροί σήμερα. Εγώ προσωπικά χαίρομαι που ακούω αυτές τις νέες προτάσεις και πιστεύω ότι τα προβλήματα που συνεχίζουν και παραμένουν στον τομέα αυτό και εδώ ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Γκοζές και ζητώ από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν υπόψη τους σοβαρά τις σημερινές μας προτάσεις, να μην δημιουργήσουν ένα νέο μονοπόλιο στην αξιολόγηση αντικαθιστώντας το λιγοπόλιο το σημερινό από μία και μοναδική δημόσια αρχή επιχείρησης. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σουίλεμπεργκ, εκ μέρους των συντηρητικών, για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε έγινε σαφές από τη χρηματοπιστωτική αγορά ότι οι οίκοι αξιολόγησης ε, έκαναν πολλά λάθη η επικαιροποίηση της ε, οδηγίας, κοινωνικής οδηγίας θα είναι πολύ χρήσιμη προκειμένου να παρακολουθούμε καλύτερα τις δραστηριότητε τους. Οι οίκοι αξιολόγηση είναι εξαιρετικά ισχυρές οργανώσεις εταιρείε και έχουν τη δυνατότητα να ε, επηρεάζουν πάρα πολύ τις αγορές. Συνεπώς θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία τους ε, συνεχώς. Όμως ε, δεν θα πρέπει να εκπλήσονται οι αγορές. Δηλαδή, οι οίκοι αξιολόγηση θα πρέπει να δημοσιεύουν τα σενάρια και τις αναλύσεις τους έτσι ώστε να ε, αυξάνουν τη διαφάνεια στην αγορά. Ε, να μην ξεχνάμε ότι η, η, η, ε, ότι το καθήκον των οίκων αξιολόγηση είναι να αξιολογούν τη φερεγγιότητα ε, και τον κίνδυνο πτώχευση ε, ακόμα και κρατών, όχι μόνο επιχειρήσεων. Δεν θα πρέπει λοιπόν να κατηγορούμε τους οίκους αξιολόγησης όταν αξιολογούν σωστά τα στοιχεία που υπάρχουν. Όμως δεν θα πρέπει βέβαια να τους επιτρέπουμε με ιδιωτελή κίνητρα να επηρεάζουν τις αγορές. Το θέμα είναι γιατί οι αγορές και τα κράτη εξαρτώνται τόσο πολύ από τους οικού αξιολόγησης αντί να κάνουν οι ίδιοι αναλύσεις και να συλλέγουν πληροφορίες γιατί μάλιστα υπάρχουν μόνο τρεις μεγάλες εταιρείες σε αυτό το τομέα. Όταν απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα τότε θα γίνει πιο σαφές πώς πρέπει να είναι υπόλογες αυτές οι εταιρείες. Thank ευχαριστώ πολύ, κυρία Σένμπερν. Ο κύριος Κλούτ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πενθυμίσω ότι χτες το βράδυ, για άλλη μια φορά, υποβαθμίστηκε από την Μούντις η Ελλάδα. Και όλοι θυμόμαστε, όλοι ξέρουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση τις τελευταίες εβδομάδες έχει ασκήσει τεράστια πίεση στους πολίτες της, στο λαό της, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο δάνειο το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα της δώσει. Το θέμα λοιπόν είναι ότι παρόλες αυτές τις προσπάθειες υποβαθμίστηκε για άλλη μια φορά η Ελλάδα και το ίδιο θα γίνει και έγινε με την Ισπανία. Μας δώσατε μια εικόνα όσον αφορά το ποιος φταίει για την υποβάθμιση, λέγοντας ότι όταν κάποιος έχει πυρετό δεν μπορεί να είναι υπεύθυνο το θερμόμετρο. Το θέμα όμως είναι αν αυτή η ανακοίνωση δεν έχει σαν αποτέλεσμα την επιδείνωση της ίδιας της κατάστασης της οικονομίας. Δηλαδή το γεγονός ότι ο ασθενής ε, διαπιστώσει ότι έχει υψηλό πυρετό μπορεί να επιδεινώσει την κατάστασή του. Ξέρετε λοιπόν ότι αυτοί οι οργανισμοί αξιολόγησης ε, αξιολογούν βάσει πραγματικών δεδομένων, αλλά πολλές φορές βλέπουμε ότι ο αντίκτυπος αυτών που κάνουν και η στιγμή που, τα την ανακοινώνουν την αξιολόγησή τους παίζει καθοριστική... καθοριστικό ρόλο και έχει τεράστια σημασία στην πτώχευση των Lehman Brothers η αντίδραση ήταν θα έλεγα έγκαιρη, επίγουσα και είχε θετικές επιπτώσεις για την συνέχεια αυτής της οικονομικής κρίσης. Για να ξεπεραστεί η σημερινή κρίση, οι οργανισμοί αξιολόγησης δεν έχουν παίξει θετικό ρόλο. Καθότι μέχρι τώρα ανησυχούμε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ανησυχούν Υπάρχει δυσπιστία όσον αφορά τα πακέτα μέτρων. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Έχετε ξεπεράσει το χρόνο ομιλία σα. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ήταν σαφή αυτά που είπα. Θα ήθελα τελειώνοντα να πω ότι οι οργανισμοί αξιολόγηση δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο έναν ιδιωτικό οργανισμό και ένα κράτος και ότι θα πρέπει να επεξεργαστούμε το σύστημα αυτό της αξιολόγησης, τους οργανισμούς αξιολόγησης, τους κανόνες και το πώς αυτό μπορεί να διαρθρωθεί εκ νέου με νέους κανόνες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπλουμ για ένα μισή λεπτό. No. Can you me Thank you very much. Sorry about that. Επίτροπε, οι οίκοι αξιολόγηση έχουν πουλήσει το κορμί του στο διάβολο εδώ και κάποια χρόνια. Όταν ξεκίνησαν να, ε, ε προ, να αξιολογούν εταιρείε ε, των οποίων ε, η, για τις οποίες αξιολογήσεις η πληρωμή τους εξαρτόταν ε, από το αποτέλεσμα της αξιολόγησης οι αξιολογήσεις αυτών των ε, ε, ομολόγων και των ε, hedge funds άλλαξε μόνο τελευταία στιγμή. Οι... Πολλές φορές όμως η αλήθεια δεν είναι πολύ δημοφιλής. Γι' αυτό πολλές φορές μισούμε τους τις οίκους αυτούς. Μην ξεχνάμε ότι η λέξη καπούτ είναι ίδια σε όλες τις ε, ε, γλώσσες, ε, ανεξάρτητα αν είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία ή το Ενωμένο Βασίλειο. Το ερώτημα είναι ποιον θα μπορούσαν να κοροϊδέψουν ψευδείς αξιολογήσεις για τελειωμένες οικονομίες. Όταν ο λαός καταλάβει ότι έγινε ε, ε, αντικείμενο κοροϊδίας και πειραματισμού θα τα κάψουν όλα και κανείς δεν μπορεί να, να τους κατηγορήσει. Ευχαριστώ κυρία Λεπέν. Για δύο λεπτά κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε επίτροποι. Δεν πρέπει να αποδείξει κανείς πλέον την αρνητική συνέπεια της δράσης αυτών των οργανισμών αξιολόγησης. Ότι ουσιαστικά ρίχνουν λάδι στη φωτιά εν μέσω της κρίσης. Και για άλλη μια φορά είδαμε ότι αναγκάζονται επιγόντως να δράσουν οι δημόσιες αρχές των ευρωπαϊκών κρατών. Οι αρχές της αγοράς, με τα διαπλεκόμενα συμφέροντα, μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λειτουργεί με σοβιετικό τρόπο δεν μπορούν παρά να δείξουν την ανηπορία τους. Ο κύριος Μπαρόζο μας είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει επιτήρηση των οργανισμών αξιολόγηση από την Κεντρική Τράπεζα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι δυνατόν να το πιστέψουμε ιδιαίτερα μετά την δήλωση του Φεβρουαρίου φέτος του κύριου Τρισέ που λέει ότι η προσπάθεια απογείωσης των ισολογισμών των τραπέζων απαιτεί εχεμήθεια, με λίγα λόγια, έλλειψη διαφάνειας και απόρριτο. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες και όχι τις αιτίε αυτής της κρίσης. Ποιος πρέπει να πληρώσει αυτούς τους οργανισμούς αξιολόγησης, αυτοί που αξιολογούνται ή αυτοί οι οποίοι θα συνεισφέρουν στον δανεισμό των ε, κρατών την ίδια ώρα βλέπουμε ότι αυτοί οι οποίοι συνεχίζουν να πολλούν χωρίς να κατέχουν και να αγοράζουν χωρίς να ε, πληρώνουν θα συνεχίσουν να είναι αυτοί που καθορίζουν τους κανόνες της οικονομίας όπως έλεγε ο Μωρίς Αλέ. Χωρίς λοιπόν κανένα αντιστάθμισμα πραγματικό θα συνεχίσει η κερδοσκοπία, η παράλογη κερδοσκοπία των χρηματαγορών και οι οργανισμοί αξιολόγησης δεν έχουν πλέον κανένα λόγο ύπαρξης. Merci. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σικρούνα για δύο λεπτά είναι ο επόμενος ομιλητής. Η πρόσφατη επίθεση των Ευρωπαίων ηγετών εναντίον των οίκων αξιολόγηση σε σχέση με το timing και το μέτρο της μείωσης της πιστολιτικής ικανότητας ε, μπορεί να θεωρηθεί από κάποιους, μπορεί να από κάποιους υπερβολικές. Ε, αλλά ο ρόλος των οίκων αξιολόγηση είναι γνωστός και όλοι συμφωνούμε ε, γι' αυτόν. Ε, οι οίκοι έχουν δώσει υψηλή αξιολόγηση ε, σε αξίες ε, που αργότερα ε, πτώχευσαν, μηδενίστηκε η αξία τους. Ε, και ε, τώρα δείχνει να είναι ένοχη αυτή η οίκη για το ακριβώ αντίθετο σε σχέση με την Ελλάδα. Ούτε το πακέτο των 750 δισεκατομμύρων δεν τους έπεισε. Ε, όμως ε, δεν θα πρέπει να φανεί ότι πυροβολούμε τον αγγελιοφόρο επειδή φέρνει κακά νέα. Η επίδραση των οίκων αξιολόγηση παγκόσμιες αγορές είναι τεράστιες. Είτε λειτουργούν σωστά είτε λειτουργούν λαθασμένα. Μπορούν να κρατούν ομήρους τις χώρες και τους κατοίκους τους. Αυτό έχει πολιτικές επιπτώσεις τεράστιες και θα πρέπει να τις αξιολογήσουμε. Θα πρέπει να δούμε πώς ε, καταλήγουν στις αξιολογήσεις τους και πώς τις πουλούν. Θα πρέπει να εξετάσουμε την ανεξαρτησία τους και τη διαφάνειά τους. Δεύτερον, ο αριθμός των οίκων αξιολόγησης και ο ανταγωνισμός μεταξύ τους. γιατί οι οίκοι αξιολόγηση ε, να μην υπόκεινται σε παρόμοιε ρυθμίσει με αυτέ τι οποίε υπόκεινται οι τράπεζε και γενικότερα ο χρηματοπιστωτικό τομέα. Οι αιτίε του προβλήματο, μεταξύ των οποίων και η σύγκρουση συμφερόντων, είναι σαφή. Η λύση δεν είναι τόσο σαφή. Συνεπώ, α προσπαθήσουμε να είμαστε αμερόληπτοι και α προσπαθήσουμε να βρούμε μια χρυσή τομή, έτσι ώστε να μην υπερβάλλουμε στην αντίδρασή μα, η οποία επίση μπορεί να έχει αρνητικέ επιπτώσει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκυκλούνα. Ο κύριο Κλίντ. Κύριε Πρόεδρε, οι οργανισμοί αξιολόγησης έχουν παίξει ένα σημαντικό ρόλο στις πρόσφατες εξελίξεις και εν μέσω της οικονομικής κρίσης. Η χρηματοδότηση, η παραγγελία αξιολογήσεων από κάποιους οι οποίοι έχουν συμφέροντα στην συγκεκριμένη δανειοδοτική διαδικασία δημιούργησε ερωτηματικά και προβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό είναι το θετικό, έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει το θέμα με πιο δυναμικό τρόπο. Θέλει να δημιουργηθεί μια ανεξάρτητη αρχή επιτήρησης, ανεξάρτητη από άποψη οικονομική, υπομορφή ιδρύματος, να μην εξαρτάται ούτε από τα κράτη-μέλη, ούτε από την Επιτροπή. Αυτή η ανεξάρτητη μορφή αυτό το Ίδρυμα μπορεί να εποπτεύσει και να ελέγξει τους τρεις οργανισμούς αξιολόγησης που υπάρχουν σήμερα και λειτουργούν σαν ένα ολιγοπόλιο. Και θα μπορεί στην περίπτωση αυτή να υπάρχουν κάθε φορά δύο αξιολογήσεις. Η μία εκ των οποίων να προέρχεται από αυτήν την Ευρωπαϊκή Αρχή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογούν αυτές τις ε, αιτήσει και κατόπιν να υπάρχει η χρηματοδότηση από τους αρμόδιους οργανισμούς. Πιστεύω ότι αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να δούμε, και αυτό καλούμαστε να κάνουμε τώρα, αν θα πρέπει να περιοριστεί λίγο η δράση αυτών των οργανισμών αξιολόγησης. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Φόρτ για ένα λεπτό έχει το λόγο. Thank you. Um, Καλωσορίζω τη συζήτηση αυτή. Είναι χρήσιμη. Θα πρέπει να δούμε την αξία των αξιολογήσεων και πώς θα ενθαρρύνουμε περισσότερες, περισσότερες οίκους για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα. Επίσης θα πρέπει να καταπολεμήσουμε το σύγκρουση συμφερόντων ε, σε ό,τι αφορά τις πληρωμένες ε, ή παραγγελμένες αξιολογήσεις. Όμως ε, αυτό το αυτή η σύγκρουση, η περίπτωση σύγκρουση ε, ε, συμφερόντων υπήρχε από παλιά και θα έπρεπε να το ξέρουμε. Επίση, για να πετύχουμε του στόχου του 2020, η Ευρώπη χρειάζεται επενδύσει και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται ε, εμπιστοσύνη στην αγορά. Οι οίκοι αξιολόγηση αποτελούν τμήμα αυτή τη εμπιστοσύνη στην αγορά. Όταν λειτουργούν σωστά, αυξάνουν την πρόσφυγη την ε, πρόσβαση ε, των ε, αγορών σε δάνεια και σίγουρα εξοικονομούν χρήματα στους φορολογούμενους ενώ ταυτόχρονα δίνουν στους επενδυτές και κάποιες κατευθυντές γραμμές. Ας θυμηθούμε ότι κανένας εκδότης 3α στην Ευρώπη δεν έχει πτωχεύσει ποτέ. Άλλωστε είναι μικρότερο του 0,3% το ποσοστό ε, πτώχευσης ε, των 3α ε, εταιριών. Από τις χώρες καμία δεν έχει πτωχεύσει από αυτές που είχε 3α. βέβαια, οπότε δεν τα έχουν κάνει και όλα λάθος, έτσι, ορισμένα λάθη έχουν κάνει. Ευχαριστώ κύριο Μοργκάντη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε συνάδελφοι, είμαι πεπισμένο ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε και την διαφάνεια και τον τρόπο με τον οποίο είναι υπόλογοι οι οργανισμοί αυτοί. Όμως δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσαμε να περιορίσουμε τη λειτουργία και το πεδίο, ε, το πεδίο λειτουργίας αυτών των οργανισμών. Εάν δεν υπήρχαν οι οργανισμοί αυτοί αξιολόγηση, θα είχαμε πολύ περισσότερες ε, χρεοκοπίε όλων των χρηματοπιστωτικών ε, ιδρυμάτων. Εγώ πιστεύω στην δημόσια αγορά και στην ελεύθερη αγορά. Άρα πιστεύω και στην λειτουργία των οργανισμών αξιολόγηση λειτουργικής ικανότητα. Μία ένα, ένα, η δημιουργία όμως ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αξιολόγησης θα ήταν ένας τρόπος χειραγώγησης της αγοράς. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι η ευθύνη τελικά αυτών των οργανισμών αξιολόγησης στην παρούσα κρίση τα δεδομένα και τα μέτρα τα οποία έχουν υιοθετηθεί, δείχνουν πως ε, κάποια κράτη στην Ευρώπη θέλησαν να αντικαταστήσουν την πραγματική οικονομία με μια, με την, ε, με τα απλά, με μια απλή δημοσιονομική ρύθμιση. Κύριε Ποδηματά, έχετε τρία λεπτά. Κύριε Επίτροπε, η σημερινή συζήτηση για το πλαίσιο εποπτείας και ελέγχου της ε, λειτουργίας των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας καθίσταται δυστυχώς ακόμα περισσότερο επίκαιρη μετά τη χθεσινή απόφαση του οίκου να υποβιβάσει κατά τέσσερις ολόκληρες μονάδες την πιστοληπτική ικανότητα της ελλάδας. δεν είναι βεβαίως η πρώτη φορά στην περίοδο των τελευταίων μηνών που η πιστοληπτική ικανότητα της ελλάδας υποβαθμίζεται σημαντικά η χθεσινή όμως υποβάθμιση είναι εξόφθαλμα προκλητική και αναιτιολόγητη καθώς δεν λαμβάνει υπόψη ούτε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή του προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης την οποία χαιρέτησαν οι εκπρόσωποι της τρόικας που βρίσκονται από χθες στην αθήνα ούτε τη δημιουργία του ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας ούτε καν το γεγονός ότι έχουν δεσμευτεί εκατόν δέκα δισεκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση των αναγκών της ελληνικής οικονομίας. είναι λογικό κύριε επίτροπε την ώρα που ο πρόεδρος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας ο επικεφαλής της deutsche bank αλλά και ο εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής επιτροπής συγχαίρουν την ελληνική κυβέρνηση για την πορεία υλοποίησης του μνημονίου συμβάλλοντας έτσι στην ανάκαμψη του ευρώ έναντι του δολαρίου αλλά και στην ανάκαμψη των ευρωπαϊκών χρηματαγορών η moody's να υποβαθμίζει περαιτέρω την ελλάδα προβαίνοντας στην εντελώς αντίθετη εκτίμηση. είναι προφανές νομίζω ότι αυτή η κίνηση αναδεικνύει ακριβώς τη σύγκρουση συμφερόντων καθώς δεν υπονομεύει απλώς τις προσπάθειες της ελλάδας για δημοσιονομική εξυγίανση αλλά δίνει το έναυσμα για να συνεχιστούν οι κερδοσκοπικές επιθέσεις των αγορών σε βάρος της ελληνικής οικονομίας αλλά και συνολικά της ζώνης του ευρώ. επιβεβαιώνεται έτσι για άλλη μια φορά ότι οι οίκοι αυτοί αξιολογούν χωρίς να διασφαλίζεται η αξιοπιστία τους και χωρίς να ελέγχονται τα κίνητρα και τα αποτελέσματα των αξιολογήσεών τους εγείροντας σοβαρά ζητήματα δημοκρατίας αλλά και κυριαρχίας εθνικής και ευρωπαϊκής καθώς μιλάμε για την αξιολόγηση οικονομιών της ζώνης του ευρώ θα μπορούσε κανεί να αναφέρει πολλά ακόμα παραδείγματα το ζητούμενο ωστόσο είναι τι κάνουμε για να θωρακίσουμε τι ευρωπαϊκέ οικονομίε από την κερδοσκοπία που προκαλούν οι αμφιλεγόμενε και αδιαφανεί αυτέ αξιολογήσει. χρειάζονται άμεσα δράσει σε δύο επίπεδα το πρώτο είναι η δρομολόγηση τη δημιουργία ενό ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού οίκου αξιολόγηση και το δεύτερο είναι η συγκρότηση ενό αυστηρού και αξιόπιστου πλαισίου λειτουργία των οίκων αυτών ενός πλαισίου λειτουργίας που θα θέτει διαφανή και ενιαία πρότυπα για τα κριτήρια αξιολόγησης για το χρόνο δημοσιοποίησης της αξιολόγησης σε συνάρτηση με την αντίδραση που προκαλείται στις αγορές και τέλος για την αξιολόγηση της αξιολόγησης σε βάθος χρόνου ως προς την ακρίβεια και την αξιοπιστία της. ευχαριστώ. ο Συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Οι οργανισμοί πιστολεπτικής, αξιολόγησης πιστολεπτικής ικανότητας, λαμβάνοντας υπόψη και όλη αυτή την κρίση, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σαν παράγοντες και αυτοί που οδήγησαν στην κρίση. Γιατί πιστεύουμε ότι οι αξιολογήσεις τους επιδίνωσαν την ε, γενικότερη κατάσταση και υποβάθμισαν την πιστοληπτική ικανότητα των κρατών και, θα πρέπει, και προφανώς δεν συνεισέφεραν στην δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης στις αγορές. Η νέα διαδικασία η οποία προτείνεται προβλέπει καλύτερη εποπτεία και διαφάνεια μεν, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να, να υπάρχει εκτός από την ε, εποπτεία αλλά και η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων σε αυτούς τους οργανισμούς αξιολόγησης. Ίσως έπρεπε να δηλαδή, ενθαρρύνουμε και τον ανταγωνισμό σε αυτόν τον, οργανισμό, σε τον, τον τομέα των οργανισμών αξιολόγηση ψηλωτική ικανότητα. Οι επόμενοι ομιλητέ έχουν ένα λεπτό μόνο στη διάθεσή του. Ο επόμενο ομιλητή ο κ. Καρά. Κύριε Πρόεδρε, η απόφαση της Μούντι δείχνει τον κυρίαρχο ρόλο στις χρηματαγοράς των οργανισμών αξιολόγησης, καθώς και την έλλειψη διαφάνειας αυτών των διαδικασιών. Θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να ελεγχθούν. Η ανεξαρτησία των οργανισμών αξιολόγησης θα πρέπει να διασφαλιστεί και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρχουν μετακινήσεις ποσών, διαπλεκόμενα συμφέροντα, συγκρουόμενα συμφέροντα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αφήσουμε αυτές τις μη διαφανείς διαδικασίες να επηρεάζουν τις οικονομίες μας. Υπάρχει σήμερα μια μονοπωλιακή κατάσταση όσον αφορά την αξιολόγηση και έλλειψη ανταγωνισμού. Χρειαζόμαστε για να αλλάξει η κατάσταση οργανισμούς αξιολόγησης που να έχουν την έδρα τους στην Ευρώπη. Ακούστηκε η πρόταση για μια τέτοια αρχή, ένα τέτοιον οργανισμό που θα λειτουργεί με μορφή ιδρύματος. Πιστεύω ότι οι προτάσεις αυτές θα πρέπει σοβαρά να εξεταστούν από την Επιτροπή. Ο κύριος Κούτες είναι ο επόμενος ομιλητής. Οι δραστηριότητες των οίκων αξιολόγησης ε, δημιούργησαν την δημοσιονομική κρίση Επιπλέον, οι αξιολογηση την επιδίνωσαν. Ο κανονισμός του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου ήταν μια προσπάθεια ρύθμιση των δραστηριοτήτων τους. Πρέπει όλοι οι αξιολογήσεις που έχουν έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να σέβονται συγκεκριμένους κανόνες, να αποφεύγουν τη σύγκρουση συμφερόντων, να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια στη λειτουργία τους και κυρίως Πρέπει να σταματήσουμε να δεχόμαστε αυτή την κατάσταση, ε, αυτή την ολιγοπολιακή κατάσταση. Δεν είναι δυνατόν η αγορά να επηρεάζεται από τη βαθμολόγηση τριών αμερικανικών οίκων. Ο, όταν ένα κράτος ε, πτωχεύει, δεν είναι δυνατόν ε, τα επίσης και αξιολόγησης να του, επί, να του απαγορεύουν να δανειστεί. Ο κύριος Μέλτες, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, είναι τελείως παράλογο να αποφανθεί μόνον ένας οργανισμός αμερικανικός και ιδιωτικός για ένα θέμα που αφορά ένα ολόκληρο κράτος, ένα δημόσιο έλλειμμα. Πρέπει λοιπόν εδώ να δημιουργήσουμε μία διαφορετική κατάσταση στην Ευρώπη με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και όσον αφορά τις αξίες και όσον αφορά τα ομόλογα, τα χρεόγραφα και όλες τις άλλες κατηγορίες αξιών που αξιολογούνται. Εδώ υπάρχει μια τεράστια πίεση από μέρους των Αμερικανικών αυτών οργανισμών και η ποιότητα, αν θέλετε, αυτών των οργανισμών αξιολόγησης πολλές φορές αμφισβητείται. Βλέπουμε ότι σήμερα σε αυτή την ε, οικονομική κρίση θα πρέπει να περιοριστεί ο ρόλος των ε, οργανισμών αξιολόγησης, οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να μην βρίσκονται καθόλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πάντα να έχουν την έδρα τους εκτός. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κύριε, κύριε Πρόεδρε, μέσα στα πλαίσια της παρούσας κρίσης, ο ρόλος των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αμφισβητείται όλο ένα και περισσότερο, διότι από ό,τι φαίνεται... Ε, δεν μπόρεσαν αντικειμενικά να αξιολογήσουν την ε, πιστοληπτική ικανότητα όχι μόνο ε, ιδιωτικών εταιριών, ε, ιδιωτικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά και κρατών. Και υποβάθμισαν κάποιες την πιστοληπτική ικανότητα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιδίνωσαν την οικονομική κρίση τρεις ε, ούτως ή άλλως, ε, ε, τρεις, τρεις είναι οι οργανισμοί αξιολόγησης, αμερικανικοί οργανισμοί οι οποίοι ελέγχουν όλη την αγορά. Υποστηρίζω την πρόταση του κύριου Μπαρόζο να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός οργανισμός. Ξέρετε ότι την προηγούμενη εβδομάδα ένας από τους οργανισμούς υποβάθμι, άλλαξε τη βαθμολογία της, της Γερμανίας μετά από ένα, από ένα λάθος. Ο λόγος του Στρέιτσεκ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, άκουσα προσεκτικά την συζήτηση που λαμβάνει η χώρα εδώ. Εγώ ε, δεν είμαι υπερασπιστής ε, των οίκων Δεν εκφράζω τα συμφέροντά τους επουδενή, αλλά από την άλλη μεριά δεν φοβούμαι ή δεν διστάζω να δω και τα θετικά τους. Ασφαλώς και δεν μ' αρέσουν οι ολιγοπολιακές ή μονοπολιακές καταστάσεις. Το ερώτημα όμως είναι γιατί πολλές χώρες έπεσαν τόσο βαθιά σε δημοσιονομική κρίση. Ενδεχομένως διότι το κράτος παρεμβαίνει πάρα πολύ στην ελεύθερη αγορά. Λοιπόν, αν συζητούσαμε αυτά τα πράγματα, θα συζητούσαμε για λιγότερο χρόνο ε, το, το, θέμα των οίκων αξιολόγηση. Κυρία Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για την δώσετε τη δυνατότητα να παρέμβω σε αυτή τη συζήτηση λίγες μέρες μετά την υποβάθμιση ε, τον, της Ελλάδας από, μια, από έναν τέτοιο οργανισμό αξιολόγησης πολιτικής ικανότητας. Έχω την εντύπωση ότι ο ρόλος αυτός, ο ρόλος τους, ο ρόλος των οργανισμών έχει δεσμοθετηθεί. Ε, ρυθμίζουν με το ρόλο τους την ε, πολιτική κατάσταση. Επηρεάζουν την, την οικονομική κατάσταση της, της Ευρώπης, επιδεινώνουν την οικονομική κρίση, ε, υποβαθμίζουν ε, τα κρατικά ομόλογα, τα δημόσια χρέη των χωρών και θα πρέπει οι οργανισμοί αυτοί να λειτουργούν με διαφάνεια και με κοινά πρότυπα. Διότι τα λάθη τους, τα λάθη τους μπορεί ή να, οδηγήσουν στη χρεοκοπία μιας επιχείρησης ή να επιδεινώσουν ακόμα περισσότερο ε, μια, οικονομική κρίση. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να, γίνουν δημόσιοι οργανισμοί αυτοί, όμως θα πρέπει να μπορούν να είναι υπόλογοι οργανισμοί αυτοί απέναντι στι κυβερνήσει. και πιστεύω θα πρέπει να βρεθεί μια σωστή ισορροπία για να εξασφαλίσουμε και ένα ευρωπαϊκό μέλλον. Ο κύριο παπα Παπα-Νικολάου. Κύριε Επίτροπε, κυρίε και κύριοι, πράγματι εγείρει πολλά ερωτηματικά η χθεσινή υποβάθμιση τη πιστοληπτική ικανότητα τη Ελλάδα από τον Νίκο Μούντι. αναφέρθηκε και από του συναδέλφου. Προσθέτω εδώ ότι στι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική και για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε το πλαίσιο λειτουργία αυτών των οίκων αν τελικά είναι καθαρό αν είναι διαφανέ αν είναι θεσμοθετημένο. οι περισσότερε λοιπόν προσφυγέ ιδιωτών στη ηπα κατά των συγκεκριμένων εταιριών δεν δικαιώνονται λόγω ενό νόμου του 1933, που ορίζει πω οργανισμοί αξιολόγηση δεν έχουν ευθύνη για τα ποσά που χάνονται εξαιτία λάθο εκτιμήσεών του. η δράση λοιπόν των συγκεκριμένων οργανισμών τείνει να γίνει ανεξέλεγκτη. το κερδοσκοπικό παιχνίδι δεν έχει όρια δεν έχει σύνορα και η απουσία ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου βάζει την ευρωπαϊκή ένωση όλε τι χώρε σε μεγάλε περιπέτειε. οφείλουμε να αντιληφθούμε ότι ελεύθερη οικονομία δεν σημαίνει νόμο τη ζούγκλα. οφείλουμε να αντιληφθούμε ότι δεν σημαίνει ασυδοσία. και όπου αυτό δεν γίνεται αντιληπτό κατανοητό αυτό πρέπει εμεί να το απαντήσουμε με την νομοθεσία μα να το επιβάλλουμε με τον νόμο. είπατε κύριε επίτροπε πιο ανταγωνιστική πιο πολυάριθμη οίκη. Περιμένουμε πολλά από την Επιτροπή το προσεχές διάστημα. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, ακούσατε ερωτήσεις, επιχειρήματα και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ όλες και όλους για την ποιότητα των παρεμβάσεών σας και την ειλικρίνειά σας. Δεν θα επανέλθω στο ρόλο των οίκων αξιολόγηση και, και στην σημασία των αξιολογήσεων του, Η κυρία Κόμη το υπενθύμησε πολύ πρόσφατα. Δεύτερη αρχική παρατήρηση, ο κύριος ε, Παπα-Νικολάου και ο Στράσεκ ε, είπαν ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε την λειτουργία του και είναι σωστό αυτό. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια Ε, θα πρέπει οι του να είναι όσο πιο αντικειμενικέ και αμερόληπτες γίνεται και θα πρέπει να το πετύχουμε αυτό. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως οι χρηματοπιστωτικές και άλλες εταιρείε δεν θα πρέπει να τη χάνουν σωστής και υγιού διαχείρισης. Και τα κράτη επίσης θα εξακολουθήσουν να πρέπει να διαχειρίζονται σωστά τα οικονομικά τους. Τώρα, επανέρχομαι στου οίκου αξιολόγηση. Η καινούργια πρόταση τροπή του κανονισμού που διέπει αυτού του οίκου θέλουμε να υιοθετηθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλιστεί καλύτερη εποπτεία του από την ΕΣΜΑ. Κυρία Λεπέν, Α διορθώσετε λίγο τι πληροφορίε σα. Ούτε η Ευρωπαϊκή Εντική Τράπεζα, ούτε η Κομισιόν θα αναλάβουν την εποπτεία αυτών των οίκων. Ε, εμείς θέλουμε και είναι λογικό η καινούργια αυτή ανεξάρτητη αρχή η ΕΣΜΑ να αναλάβει την εποπτεία τους για να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά που ασφαλώς είναι απαραίτητη. Αυτό το καταλαβαίνουμε βλέποντας τα όσα συνέβησαν τα τελευταία χρόνια. Όπως είπα και στην αρχή τη προηγούμενη παρεμβασή μου, αυτέ οι προτάσει και το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα πρέπει να εφαρμοστεί σωστά από τώρα μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι ε, μάλιστα ε, ε, αυτά, αυτά τα δύο και οι προτάσεις και, η, και, ισχύουσα, και το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο δεν λύνουν όλα τα προβλήματα. Για παράδειγμα, η αύξηση του ανταγωνισμού, η διαφοροποίηση. Πολύ συνάδελφοι ότι δεν θα πρέπει και αξιολόγηση να είναι λίγη. Ε, επίσης, το μοντέλο του, ε, του εκδίδοντος που πληρώνει την αξιολόγηση. Ε, είναι βιώσιμο αυτό το μοντέλο. Πρέπει να το αναρωτηθούμε. Ο κύριος Κάρας επίσης αναρωτήθηκε για αυτό το θέμα. Θα πρέπει να το εξετάσουμε αξιολογώντας τους κανόνες της καινούριας νομοθεσίες που θα τεθεί σε εφαρμογή μέχρι το Δεκέμβρη του τρέχοντος έτους. Πρέπει να εντοπίσουμε τις συγκρούσεις συμφερόντων για να τις μειώσουμε. Θα δούμε αν αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο θα είναι επαρκές ή όχι. Τρίτο θέμα που θα πρέπει να εξετάσουμε η εθνική και κοινωτική νομοθεσία. Μήπως και οι δύο βασίζονται υπερβολικά την στις των οίκων. Εγώ αυτό πιστεύω. Και τέλος, η ειδική μεθοδολογία που θα πρέπει να ακολουθείτε για το δημόσιο χρέος. Ευχαριστώ τον κύριο Πλελέντο που υποστήριξε την, τον γρήγορο συμβασμό για το πακέτο που έχουμε υποβάλει, γιατί πραγματικά την αίσθημα τη χρειαζόμαστε. Το συντομότερο δυνατό. Ασφαλώς χρειαζόμαστε μια απάντηση πιο διαρθρωτική, πιο δομική. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε και προβληματιζόμαστε για τα προηγούμενα θέματα που σας εξέθεσα. Επίσης για την ανεξαρτησία τους. Την ανεξαρτησία των οίκων προκειμένου να εξασφαλίσει η αξιοπιστία τους. Και θέλουμε ασφαλώς να εξασφαλίσουμε επίση τον ανταγωνισμό και ενδεχομένω θα έπρεπε να δημιουργήσουμε και ένα ευρωπαϊκό οίκο αξιολόγηση, ειδικά ίσω για το, για το δημόσιο χρέο. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε αυτό, αυτός ο ευρωπαϊκό οίκο να είναι κρατικό, ιδιωτικό, ε, ε, μάλλον δημόσιο, ε, ιδιωτικό ή μεικτή φύσεως. ίσως θα έπρεπε να είναι ένα ίδρυμα. Το εξετάζουμε. Θα το εξετάσουμε τις επόμενες εβδομάδες. Κυρία Μπόλση, Κάποιοι άλλοι, η κυρία Ποδηματά επίσης, αναφέρθηκαν ε, στην ε, πρόσφατη υποβάθμιση της Ελλάδας. Εγώ δεν θα ήθελα ως επίτροπος να σχολιάσω, να αρχίσω να σχολιάζω λεπτομερώς την κάθε βαθμολόγηση ε, κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα, διότι και οποιοδήποτε σχόλιο δεν θα άλλαζε τη γνώμη μας για τις αξιολογήσεις. Όμως, όπως είπε και ο συνάδελφος μου όλοι η Ρέν εδώ σήμερα το πρωί, θέλω να εκφράσω την έκπληξή μου από, για το timing, ε, τη χρονική συγκυρία αυτής της υποβάθμισης που είναι χτες. Ε, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και θα πρέπει να το διαλαλήσουμε ε, τις ε, πολύ καλές προσπάθειες ε, που καταβάλει η Ελλάδα για να εξηγιάνει τα δημόσια οικονομικά της. Και η Κομισιόν εμπιστεύεται αυτές τις προσπάθειες, δεν είναι εύκολες, αλλά είναι απαραίτητες και θα πρέπει να καταλήξουν. Άλλωστε, η Ελλάδα δεν είναι μόνη της. Βρίσκεται, κινείται μέσα σε ένα πλαίσιο ευρωπαϊκής αλληλεγγύης που υιοθετήθηκε από τους αρχιούς κρατών και κυβερνήσεων, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Κομισιόν και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πριν από μερικές εβδομάδες. Αυτό το πλαίσιο θα εξακολουθήσει να ισχύει. Ε, η πρόσφατη υποβάθμιση με οθεί ακόμα περισσότερο να εργαστώ τις επόμενες εβδομάδες ε, σε συνέχεια της ανακοίνωσής μας της Δευτέρας Ιουνίου έτσι ώστε στο τέλος του ε, χρόνου, αρχές του επόμενου έτους να έχω έτοιμες προτάσεις μας. Μην ξεχνάμε όμως ότι δεν μιλάμε μόνο για τους οίκους αξιολόγησης σε αυτή τη συζήτηση. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι ε, η αξιολόγηση είναι ένα εργαλείο γενικότερα που θα πρέπει να βελτιώσουμε μέσα στο πλαίσιο μιας γενικότερης αρχιτεκτονικής που θα βασίζεται στην αποτελεσματική εποπτεία και στην έξυπνη ρύθμιση. Και το λέω και το ξαναλέω, ε, θα πρέπει να εξάγουμε τα σωστά συμπεράσματα. Ε, θα πρέπει η επιτήρηση να αφορά όλους, προϊόντα, επιχειρήσεις, κράτη κλπ. Η ατζέντα που υπέβαλε η Κομισιόν στις 2 Ιουνίου υποστηρίζεται υποστηρίχθηκε πριν από μερικές μήνες από τους υπουργού στο Λουξεμβούργο και ελπίζω θα υποστηριχθεί και από τους αριούς κρατών κυβερνήσεων στο, Συμβούλιο, στο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα ήθελα και τη δική σας υποστήριξη έτσι ώστε σιγά σιγά να χτίσουμε το σύνολο των δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει. Σε συνεργασία με τους εταίρους μας, ιδιαίτερα στις ε, Ηνωμένες, τις υπόψη τα συμπεράσματα τα οποία έχουμε βγάλει τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Έκθεση Κλίντς δημόσια προσφορά κινητών αξιών και εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας. Ο λόγος στον εισηγητή. Τέσσερα λεπτά. Ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε,